Herr Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. η συνεδρία Τακτικά. της χθεσινές συνεδρίασης μαζί με τα έγγραφα που ενεκρίθησαν είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Εν αυτή ε, περίπτωση εγκρίνεται. Ένσταση ήταν αυτό. Όχι. Ε. Δεν είχατε αντίρρηση για τα πρακτικά. Καλώς εγκρίνονται λοιπόν. Τώρα έχουμε τη συζήτηση συστήσει περιπτώσεων παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Δυνάμει του άρθρου 122 του κανονισμού. Τι Λατσάλετ. Σαλή είναι η πρώτη υπόθεση και θα ακούσω το συναδέλφου που έχουν γραφεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 8, άνοιξα την ιστοσελίδα του Γκυλάντ Σαλίτ εδώ στο Κοινοβούλιο. Και ένα πράγμα μου έκανε ε, υπόψη. Έχουν περάσει από τότε που συνελήφθη 1351 ε, μέρες 18 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Από τότε ζει μακριά από τον πατέρα του, την αδελφή του και τη μητέρα του. Στην ίδια ιστοσελίδα διάβασα ένα κείμενο βιβλικό από τον προφήτη Ερεμία και έλεγε αστραφούμε στραφούμε προς τον Θεό και ας ζητήσουμε από τον Θεό να επιτρέψει στα τέκνα μας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ο Γκυλάτ Σαλίτ λέει ο μιλητής κοιτώντας προς τον ουρανό θα πρέπει να επιστρέψει και αυτό στη γη του Ισραήλ που είναι η πατρίδα του. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το απόγευμα συζητάμε την υπόθεση του Γκυλάτ Σαλίτ με αφορμή ε, μια συζήτηση της αντιπροσωπείας με το Ισραήλ χθες είπα ότι η απελευθέρωση του Γκυλάντ είναι δική μας υπόθεση και όχι μόνο υπόθεση των Ισραηλινών και της οικογένειάς του. Νομίζω ότι το ψήφισμά μας σήμερα το απόγευμα αυτό δείχνει ότι δηλαδή το θέμα αυτό μας απασχολεί Η περίπτωση του Γκυλάντ Σαλίτ, επαναλαμβάνω, είναι και θέμα ευρωπαϊκό, είναι θέμα όλων μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να ξαναβρει την οικογένειά του ο Γκυλάντ Σαλίτ, το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Ρίς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ο Γκυλάτ Σαλίτ ήταν 19 ετών όταν απήχθη σε μια επίθεση τη χαμά κοντά στη Γάζα. Όχι στην ίδια δηλαδή, τη Γάζα, αλλά σε ένα κυμπούτσι στο Ισραήλ. Εκεί ε, ε, βρισκόταν με, με το απόσπασμά του. Εδώ και τέσσερα χρόνια ζει σε ένα μπουντρούμι χωρίς δικαίωμα επίσκεψης, χωρίς ε, γιατρό, δικηγόρο, χωρίς αλληλογραφία, χωρίς ε, να ισχύει γι' αυτόν η σύμβαση της Γενέβης. Ενώ ο Κιλάτ Σαλίντ ασκούσε τη στρατιωτική θητεία όπως όλοι οι συνομιλικοί του. Σήμερα είναι μαζί μας ε, στην Ολομέλεια ο πατέρας του Γκυλάτ Σαλίτ. Στον Γκυλάτ ε, άρεσαν τα ε, μαθηματικά, το ποδόσφαιρο και θα ήθελε πολύ να γυρίσει αν δεν ζούσε μια τρόγλη τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποκομμένο από τον κόσμο και από την οικογένειά του. Σήμερα, κύριε Επίτροπε, δεν θέλω να μιλήσουμε για πολιτική, δεν θέλω να μιλήσουμε για τη Μέση Ανατολή, για διενέξει, συγκρούσει, ε, ανταλλαγέ κρατουμένων. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα, ομόφωνο και σύσσωμο, συζητά να επιτρέψουμε σε ένα νέο να επιστρέψει στο σπίτι του. Ένα νέο Ισραηλινό, ένα νέο Γάλλο, ένα νέο Ευρωπαίο. Γι' αυτό έστειλε επιστολή σήμερα στη Λέιδη Άστον μαζί με του συντάκτε του ψηφίσματο από έξι πολιτικέ ομάδε, την κυρία Σάγια, τον Γκάουν Μπεντίτ, Ρίτσαρτ Χάουιτ, Τάνοκ και Μπάστιαν Μπέλντερ, ζητούμε όλοι στεναρά να πάει η Βαρόνια Άστον στο Ισραήλ, που ούτως θα πάει στο Ισραήλ και στην Λωρίδα της Γάζας την επόμενη Τετάρτη να χρησιμοποιήσει ε, την έγκλη τη, το κύρο τη, όπω απορρέει και από το δικό μα ψήφισμα, το κύρο που απορρέει από την ομοποίηση 500 εκατομμυρίων πολιτών που εκπροσωπούμε σήμερα και να ζητήσει επίμονα την απελευθέρωση του κοιλάτου Σαλίτ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Δερόσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ το κοινό ψήφισμα από όλες τις ομάδες για την απελευθέρωση του Κιλάτ Σαλίτ που πήχθη από το ζωτικό σκέλο τη χαμά και ο πατέρα του μα εξήγησε χθε ότι είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και θα πρέπει να μετατραπεί σε πολιτικό ποδόσφαιρο. Δεν θα πρέπει λοιπόν ποτέ να λησμονούμε μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση πόσο υποφέρουν οι οικογένειε των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τα παιδιά του, που τα παιδιά του έχουν κρατηθεί εχμάλωτοι. Η σύμβαση τη Γενέβη πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλε τι πλευρέ. Δεν είναι αποδεκτό ότι δεν αναγνωρίζει το καθεστώ του εχμαλώτου πολέμου στον Χιλάτ Σαλίτ και ότι δεν έχει την προστασία την οποία δικαιούται δεν έχει η οικογένειά του ενημέρωση για την ε, σωματική ή ψυχολογική του υγεία. Επίσης, ταυτόχρονα έχουμε 7.200 Παλαιστινίου κρατουμένου στι Ισραηλινές φυλακές, πάλι με παραβίαση των συνθήκων της Σύμβαση τη Γενέβη, εκ των οποίων πολλοί ε, έχουν ήδη εκτίσει πάνω από 25 χρόνια φυλάκιση. Από αυτού είναι πολλά τα παιδιά. Από αυτού είναι και πολλά τα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου που κρατούνται μόνο και μόνο σε αντίπεινα για την ε, κράτηση του Χιλάτ Σαλίτ. Έτσι λοιπόν, και μια και θα πάω στην Ιορδανία με την Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη αυτήν την εβδομάδα, θα ήθελα να πιέσουμε όπως και η Λέιδη Άστον ε, τους Ισραηλινούς και την Χαμάς. Τη Χαμάς να απελευθερώσει τον Χιλάτ Τσαλίτ και, τον, και, τους, και τους Ισραηλινούς να απελευθερώσουν τα παιδιά που βρίσκονται φυλακισμένα στις φυλακές τους. Ευχαριστώ κύριε Τερόσα. Κύριο Στάνοκ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ο Λοχίας Σαλίτ ε, βρίσκεται κρατούμενος Χαμάς εδώ και τρία χρόνια. Ε, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι είναι εχμάλωτος πολέμου. Όμως ε, το Ισραήλ και σωστά πιστεύω, λέει ότι απλώς είναι θύμα απαγωγής. Βρίσκεται κρατούμενο στη Γάζα, δεν έχει καμιά επαφή και επικοινωνία με τον έξω κόσμο, δεν έχει καν ε, πρόσβαση η Διεθνής ε, Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στον κρατούμενο αυτό. Η οικογένειά του μόνο ένα βίντεο έχει δει ε, με στοιχεία από τη Χαμάς που δείχνουν ότι ήταν ζωντανός, αλλά άλλα στοιχεία για την ε, κατάστασή του δεν έχει λάβει. Έτσι λοιπόν, αν θέλει η Χαμά να τη σοβαρά υπόψη από τη διεθνή κοινότητα, θα πρέπει να βελτιώσει άμεσα τι συνθήκε κράτησή του με βάση για τον ανθρωπιστικό διεθνέ δίκαιο. Αλλά δεν μα αρκεί εμά αυτό. Εμεί θέλουμε άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση του Σιλάτ Σαρίτ. Εγώ ξέρετε ότι ποτέ δεν υποστηρίζω την, ε, το διάλογο με την τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμά. Εάν ε, πρόκειται να αναπτύξουμε διάλογο, το μόνο αντικείμενο διαλόγου θα πρέπει να είναι η απελευθέρωση του Χιλάτ Σαλίτ. Ευχαριστώ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνήθω όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει ψήφισμα, ε, ειδικά για τη Μέση Ανατολή, είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε και να υπάρχει σύμπνοια. Στην περίπτωση αυτή υπήρξε ομοφωνία χάρη στου συναδέλφου που συνέταξαν το ψήφισμα. Η κατάσταση του του Σαλίτ είναι ανθρωπιστικό ζήτημα. Και αυτό υπογραμμίζει και το ψήφισμά μα, ότι από τη στιγμή που εχμαλωτίστηκε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, κρατείται σε άγνωστο μέρο, στη Γάζα, και στερείται τα στοιχειώδη δικαιώματα ε, και καμία ανθρωπιστική ε, προδιαγραφή. Καταπατάται και το άρθρο 3 της Συνθήκης της Γενέβης. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση του Τζιλάτ Σαλίτ και το ελάχιστο, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι οι γονείς του και ο Ερθρός Σταυρός να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί του δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε την αξία μια ανθρώπινη ζωή. Δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο παζαρέματο μεταξύ τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμά και του Ισραήλ. Θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα, αμέσω. Αυτό είναι το ε, μήνυμα που θέλουμε η υπατική πρόσωπο να μεταφέρει στη Γάζα στην επόμενη τη επίσκεψη εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συναδέλφε Σάια. κύριο Χατζηγεωργίου, παρακαλώ, για δύο μισή λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, χθε ε, συμμετείχα μαζί με άλλου συναδέλφου σε μια συνάντηση στην οποία ήταν παρόν ο πατέρα του Σαλίτ και θέλω να πω ότι κανένα δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητο από το δράμα αυτή τη οικογένεια. Γι' αυτό και εμά θέση μα είναι ότι ο Γκυλάτ Σαλίτ, μέλο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθηκε μέσα στο έδαφο του Ισραήλ στι 24 Ιούνιου του 2006, πληρεί τα κριτήρια για να θεωρηθεί εχμάλωτο πολέμου σύμφωνα με την τρίτη συνθήκη τη Γενέβη. ω εκ τούτου θα πρέπει να τη χάνει ανθρώπινη μεταχείριση και να του επιτρέπεται επικοινωνία. θα πρέπει να επιτραπεί στο διεθνή ερυθρό σταυρό να τον επισκεφθεί και η οικογένεια έχει κάθε δικαίωμα να έχει ενημέρωση για την κατάστασή του καθώ βεβαίω και να τον επισκεφθεί. ταυτόχρονα εκφράζουμε την θέλησή μα την πίστη μα, αυτό ο άνθρωπο να απελευθερωθεί. Όμω, αγαπητοί συνάδελφοι χωρί να θέλω καθόλου να μειώσω όσα έχω πει μέχρι στιγμή, νομίζω ότι είναι λίγο απολύτικη η στάση μας να θεωρούμε ότι μπορεί αυτό το ζήτημα να διαχωριστεί από ένα σωρό άλλους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στις φυλακές και που είναι επίσης ανθρωπιστικό ζήτημα η παρουσία τους σε αυτές τις φυλακές. Θεωρώ μάλιστα ότι δίνουμε και φρούδες ελπίδες σε αυτή την οικογένεια αν νομίζουμε ότι εστιάζοντας σαν κοινοβούλιο στην απελευθέρωση ενός του συγκεκριμένου αυτού ανθρώπου που επαναλαμβάνω την απέτησή μας να απελευθερωθεί. Νομίζω όμως ότι δίνουμε φρούδες ελπίδες εάν εστιάζουμε την εικόνα μας μόνο προς αυτό το σημείο, θεωρώντας ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Δεν είναι ανθρωπιστικό το ζήτημα του γεγονότος ότι βρίσκονται στις φυλακές δεκάδες παιδιά Παλαιστινίων που είναι 16 χρονών. Πώς μπορείς να διαχωρίσεις αυτά τα δύο ζητήματα δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο γεγονό ότι η ίδια η γάζα επειδή αναφέρθηκε προηγουμένω ότι ζει σε μια τρόγλη και ζει σε μια τρόγλη αυτό το παιδί η ίδια η γάζα είναι μια απέραντη τρόγλη αγαπητοί συνάδελφοι. ενάμιση εκατομμύριο παλαιστίνοι που ζουν εκεί ε, ζουν μια συλλογική τιμωρία. υπάρχουν 7.200 παλαιστίνοι στι Ισραηλινέ φυλακέ, ανάμεσά του 270 παιδιά 16 18 χρόνων 44 παιδιά κάτω των 16. Από το 67 μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί και πάει στις φυλακές 750.000 Παλαιστίνοι. Απαιτούμε λοιπόν την απελευθέρωση του Σαλίτ. Είναι απολύτικη όμω τάση να θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα χωρί να διασυνδεθεί με μια συνολική εικόνα που υπάρχει στην Παλαιστίνη. Κλείνω με αυτό. Η μόνη περιοχή του κόσμου που έχει υπουργό για φυλακισμένου είναι η Παλαιστίνη. Εκφράζω ξανά την αγάπη και τη συμπάθειά μας στην οικογένεια και ελπίζω σύντομα αυτό το πρόβλημα να λυθεί. ευχαριστώ κύριε Χατζηγεωργίου. Η κυρία Κιλ Νίλσεν για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ψήφισμα για τον Λοχία 19 Κιλάρ Σαλίτ ε, αποτελεί συνέχεια μια σειρά από ψηφίσματα που είχε θετήσει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση των δικαιωμάτων στη Μέση Ανατολή. Ο Δεκανές Χιλάτ Σαλίτ είναι κρατούμενο εδώ και 1355 μέρε. Πρέπει να απελευθερωθεί αμέσω. Αυτό απαιτούμε και σε αυτό ελπίζουμε με όλη μα την ψυχή. Ο νέο δε Γάλλος, Γαλλοπαλαιστίνιος Αλάμουρη, ο οποίος βρίσκεται από τις 13 Μαρτίου του 2005 στα χέρια των Ισραηλινών πρέπει και αυτός να απελευθερωθεί. Το ίδιο και όλοι οι κρατούμενοι Παλαιστίνοι που, για τα παιδιά ιδιαίτερως που βρισκόνται κρατούμενα σε, παράβαση κάθε, σε παραβίαση κάθε είδους διεθνούς συνθήκης και κυρίως δικαιωμάτων των παιδιών. Ο Αμπταλά Ραμάτ από το Ιλμπιλίν πρέπει να απελευθερωθεί. Τα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, ο Μαρουάν Μπαρμπουτή παραδείγματι, πρέπει να απελευθερωθούν. Πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει απερίφραστα τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου στη Μέση Ανατολή. Τα ψηφίσματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την καταστολή και τη βία όπως ε, είδαμε να συμβαίνει με τη δολοφονία ενός μέλους της Χαμάς στο Ντουμπάι που ε, λυπούμαστε που έλαβε χώρα γιατί καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την, δύσκολο τον αγώνα για την απελευθέρωση του Χιλάτ Σαλίτ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τώρα ακούμε εκ μέρου των ομάδων ομιλητές. Η κυρία Μπεσέσκου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε είναι η δεύτερη φορά που λαμβάνω το λόγο στην Ολομέλεια για να μιλήσω για τον Γκυλάτ Σαλίτ. Και χαίρομαι που χάρη στι κοινέ μα προσπάθειε ε, καταλήξαμε σε αυτό το κοινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η σύμνη και ομοφωνία δείχνει την ανησυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Τα δικαιώματα του Τζιλάντ, όπω περιλαμβάνονται στην Τρίτη Σύμβαση τη Γενέβη, δεν θα πρέπει να αποτελούν όρο για την επίλυση του Ισραηλοπαλαιστινιακού ζητήματο. Άλλωστε, ο, ο πατέρα του Τζιλάντ Χαλίδη είπε ότι ούτε αυτό ούτε η οικογένειά του ε, έχουν οποιασδήποτε διασυνδέσεις με πολιτικούς ή έχουν εμπλακεί με την πολιτική. Αν θέλουμε μια ειρηνική συνύπαρξη δύο κρατών που θα συζούν με ειρήνη και ασφάλεια θα πρέπει να προβούμε σε συμφωνία και απελευθέρωση του Τζιλάτ Σαλίτ. Βέβαια ζητήθηκε η ανταλλαγή του Τζιλάτ Σαλίτ με χίλιους Παλαιστίνιου κρατούμένου. Η οικογένεια του Τζιλάτ χρειάζεται την βοήθειά μα και τη συμπαράστασή μα. Η για να... και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η υπόθεση του Τζιλάτ Σαλίτ έχει αναδειχθεί σε σύμβολο τη ματέωσης του εκνευρισμού και τη απογοήτευση, τη απόγνωση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και για όσου διαβιούν εκεί και για την παγκόσμια κοινότητα. Ο Τζιλάτ Σαλίτ είναι ένα άνθρωπο ε, το πεπρωμένο το οποίο έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ε, ενώ εφαρμόζεται το οφθαλμόν αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος δυστυχώς στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι μόνο ο Τζιλατσέλη και πολλοί άλλοι υποφέρουν στη διένεξη αυτή. Και πολύ συχνά μιλούμε για το διεθνές δίκαιο, αλλά ξεχνούμε τη στοιχειώδη επίδειξη ανθρωπιάς. Ας προσπαθήσουμε να νιώσουμε πώς αισθάνονται οι οικογένειες των θυμάτων, οι οικογένειες αυτών που υποφέρουν ή οι ίδιοι οι φυλακισμένοι. Ας απελευθερωθεί ο Τζιλατσέλιτ αφού δεν εκρεμεί δίκη εις βάρος του, ούτε έχει καταδικαστεί. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν το θάρρος να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άουκεν, παρακαλώ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση σήμερα συμβάλλει στο να βάλουμε όνομα και πρόσωπο στον ανθρώπινο πόνο και να εκφράσουμε τη συμπόνια μας στους ανθρώπους αυτούς. Είναι πολύ καλό λοιπόν το ότι μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε για τον Γιλάτ Σαλίτ ως αντικείμενο αυτού του ψηφίσματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας και στα άλλα θύματα των παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων στα δικά του δεινά, στα δεινά των οικογενειών του. Μιλήσατε και πολύ σωστά, αγαπητοί συνάδελφοι, για τι χιλιάδε των Παλαιστινίων οι οποίοι βρίσκονται κρατουμένοι σε απαράδεκτε συνθήκε κράτη, σε συνθήκε οι οποίε παραβιάζουν κάθε είδο ε, ε, κανόνα διεθνού δικαίου. Και γι' αυτό συμπάσχουμε με αυτού όπω και με τον Χιλάτ Σαλίτ και την οικογένειά του. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε αμέσως δράση και να πάψουμε να επικεντρωνόμαστε σε ένα μόνο πρόσωπο, σε ένα μόνο κρατούμενο, όταν τα θύματα αυτής της σύγκρουση είναι χιλιάδες. Υπογραμμίζω επίσης ότι απαραίτητο είναι να διερευνήσουμε τις αιτίες αυτή τη της να μην μένουμε στην επιφάνεια δηλαδή. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν πράττουμε τίποτε, εάν δεν αναλάβουμε δράση, εάν δεν ασχοληθούμε ουσιαστικά όχι μόνο με τη Γάζα, αλλά με την κατοχή τη Παλαιστίνη, εάν δεν προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτών των δύο κρατών που θα, θα θέλαμε να υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, δεν μπορούμε να δώσουμε λύσει σε αυτά τα ανθρώπινα δεινά. Πρέπει να βρούμε την καλύτερη λοιπόν λύση και ελπίζω κυρία Άστον να συμβάλλει με τη συμπεριφορά τη στην επίλυση του ζητήματο. Έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αρκείται μόνο να καταβάλει ποσά, να πληρώνει διαρκώ μόνο και μόνο για να ε, τη συνείδησή τη. Στις 25 ε, Ιουνίου του 2006, κυρίε και κύριοι, ο νεαρός δεκανέα Ατζιλάτ ε, Σαλίτ απήχθη μετά από μία τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και έκτοτε ε, κρατείται χμάλωτος, μάλιστα αποκομμένος από τον έξω κόσμο, χωρίς να έχει καμία επαφή, σε ένα σκοτεινό κελί υπόγειο και κανένας δεν μπορεί να έχει επικοινωνία μαζί του. Για, μία ακόμη φορά το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση υφίσταται την επίθεση τρομοκρατικών οργανώσεων, την επίθεση κατά του ίδιου τους του πολιτισμού. Αυτά αναφέρονται στο Ισραήλ και στην Ευρώπη. Όλοι, ο καθένας, κάθε ανθρώπινη ζωή μετράει, αλλά για τους τρομοκράτες η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει. Η Χαμάς ζητά από το Ισραήλ να ανταλλάξει χίλιους και Παλαιστίνιους εχμαλώτους συμπεριλαμβανομένων και τρομοκρατών της Χαμάς ε, σε, για να επιστρέψουν ήδη τον ε, Τζιλάτ Σαλίτ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ενδώσει το Ισραήλ σε αυτή την ανταλλαγή. Είδαμε που οδήγησαν οι ανταλλαγές ε, στο παρελθόν, πόσο τη εφορία και θριαμβευτικούς πανηγυρισμούς έχει προκαλέσει στους τρομοκράτες μια τέτοια δυσανάλογη ανταλλαγή. Δεν θα πρέπει να απαντήσει την απαγωγή του Ισραήλ με μια τέτοια ανταλλαγή κρατουμένων. Γιατί η επόμενη απαγωγή της Χαμάς μπορεί να γίνει όχι στο Ισραήλ ή στη Γάζα, αλλά στις Βρυξέλλες ή στο Άμστερνταμ. Δεν θα πρέπει να πληρώνει το Ισραήλ, αλλά η Χαμάς για την εχμαλωσία αυτή του Τζιλάτ Σαλίτ. Και το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει η Χαμάς είναι τόσο υψηλό που οικειοθελώς να τον απελευθερώσει και όχι με ανταλλαγή. Θα πρέπει να απαγορευτούν ολοσχερός όλες, ε, όλα τα ταξίδια από και προς την Ευρώπη αξιωματούχων της Χαμάς. Και αυτό θα πρέπει να ισχύσει για όλους, για όλα τα μέλη της Χαμάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ο κύριο Κέλαμ για ένα λεπτό. Ο νεαρός αυτός κρατείται για 1.400 ημέρες και φυσικά κανένα δικαίωμά του που αναγνωρίζεται από το Διεθνές Συνταγματικό Δίκαιο δεν γίνεται δεκτό. Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί νομίζω αποκλειστικά σαν ανθρώπινη τραγωδία. Υπάρχει μια τεράστια στήριξη και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν οι συνάδελφοι στον πατέρα του τραγικού στρατιώτη χτες. Είναι λοιπόν δύσκολο να πάρουμε μια απόφαση. Είναι προς το συμφέρον άλλωστε του Χαμάς εφόσον θέλουν να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή παρουσία στη διεθνή προσπάθεια για τις διαπραγματεύσεις να απολύσουν τον Σαλίτ χωρίς προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Το ψήφισμα που εξετάζουμε σήμερα δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Ούτε πρόκειται ε, να επιλύσουμε εδώ το πρόβλημα τη σύγκρουση. Απλώς θέλουμε να επιτρέψουμε σε έναν γιο να, να επιστρέψει στην οικογένεια, στον πατέρα του. Έχουμε μια οργανώση το σύνδεσμο των οικογενειών που προστατεύει και ασχολείται με, τις, με, το δράμα των Ισραηλινών και Παλαιστινίων οικογενειών που έχασαν μέλη τους σε αυτή τη διένεξη. Ο πατέρας του Τζιλάτ Σαλίτ δεν συμμετέχει σε, αυτό το, το σύνδεσμο. Έχασε όμως το παιδί του, έχει απομακρυνθεί από το παιδί του. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε με την ε, με την φράση «Ο σκοπός ε, αγιάζει τα μέσα». Δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται τρομοκρατικά μέσα για καλό σκοπό. Γιατί οργάνωση που θα προσβλέπει στο σεβασμό και την εκτίμησή μας δεν μπορεί να προσφεύγει σε απαγωγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περάσουμε στη διαδικασία Κατστιάη. Συνάδελφος Μπρέτα, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ehm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συνδέσω τη φωνή μου με όλους αυτούς οι οποίοι ζητούν να απελευθερωθεί ο Γκυλάντ Σαλίτ και εκφράζω εδώ τη συμπάθειά μου προς την οικογένεια του κρατουμένου. Κάποιοι αναρωτιόνται γιατί έχουμε ένα ψήφισμα μπροστά. Αυτό γίνεται γιατί ε, κλείνουν όπου να είναι τέσσερα χρόνια από τότε που συνελήφθη και κρατείται κάτω από απαράδεκτες, απάνθρωπες συνθήκες ο Κιλάτ Σαλίτ, όπου παραβιάζονται όλοι οι διεθνείς κανόνες και η σύμβαση της Γενέβης. Όλοι μπορούμε να γνωρίζουμε πλέον και όλοι φανταζόμαστε ότι κάθε μέρα επιπλέον κράτησης είναι μια μέρα δυστυχίας για τον Γκυλάτ Σαλίτ και την οικογένειά του. Συν της άλλης ο Γκυλάτ Σαλίτ έχει και ευρωπαϊκή υπηκότητα, είναι και Ευρωπαίος ο οποίος είναι θύμα της τρομοκρατίας και γι' αυτό ακριβώς είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέντα. Τώρα η συνάδελφος κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να καλωσορίσω εδώ την οικογένεια του Χιλάτ Σαλίτ και να τους απευθύνω φόρο τιμή για τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του. Τους υποστηρίζουμε 100%. Αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο θέλουμε να αποστείλουμε το ψήφισμα. Πιστεύουμε, όπως άλλωστε υπογραμμίζει και η έκθεση Goldtown, ότι το καθεστώς κράτησή του θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με του αχμαλώτου πολέμου. Σε αυτό έχει δικαίωμα. Όπω άλλωστε έχουν δικαίωμα και οι κρατούμενοι από τι αρχέ του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων συγκαταλαγούνται και πολλά παιδιά. Θέλουμε την απελευθέρωση όλων αυτών των κρατουμένων, και τόσο του Χιλάτ Σελίτ, όσο και των Παλαιστινίων, ανδρών, γυναικών, παιδιών. Είναι ο μόνο τρόπο αυτό να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην περιοχή αυτή. Και καλούμε την κυρία Άστον κατεπηγόντως και με όλες τις, τις δυνάμεις να πιέσει για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του Κιλάτ Σαλίτ και όλων των Παλαιστινίων εχμαλώτων πολέμου και ιδιαίτερα των νεαρών κρατουμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Κύριε Σαρνέσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το θέμα του Τζιλάτ Σαλίτ έχει μία προσωπική, μία ατομική διάσταση. Είναι η προσωπική του τραγωδία, η προσωπική τραγωδία ενός νέου ανθρώπου που είναι συνομήλικος με το γιο μου, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία οικογενειακή τραγωδία, η τραγωδία της οικογένειας του Τζιλάτ Σαλίτ. Βέβαια, έχει και πολιτικό αντίκτυπο και ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο αυτό το θέμα. Μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε η υπόθεση αυτή ότι αυτό το ασπρόμαυρο φιλμ, αυτή η ασπρόμαυρο ταινία που μερικές φορές μας παρουσιάζεται μονόπλευρα και στην περίπτωση αυτή, μια ταινία δηλαδή που μιλά για τα θύματα μόνο από παλαισθηνιακή πλευρά, είναι μάλλον ελάχιστα αντικειμενικό αυτό το φιλμ. Ζητήσαμε σήμερα ομόφωνα την άμεση απελευθέρωση του νεαρού αυτού στρατιώτη. Αλλά θα πρέπει όλοι να δείξουν υπευθυνότητα. Ευχαριστώ κύριε Σαρνέσκη. Λυπούμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Και έτσι μόνο στην συνάρφη κυρία Κορβούλα μπορώ να δώσω το λόγο προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε όλοι, το ψήφισμα το οποίο συζητάμε σήμερα αφορά ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί με αποκλειστικά ανθρωπιστικό τρόπο και όχι ε, με πολιτικό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να μην σιωπάσουμε. Έχει δημιουργηθεί μια απαράδεκτη κατάσταση. Είναι ένα θέμα εντελώς ανθρωπιστικού δικαίου θα έλεγα και θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα του κρατουμένου. Ευχαριστώ. Έχουν κατεθεί 7 προτάσεις ψηφίσματος. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει μετά το πέρας των συζητήσεων. Ζητώ συγγνώμη. Σας λησμόνησα. Πριν κλείσουμε το θέμα θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Ποτόρσνικ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η περίπτωση του Γκυλάτ Σαλίτ που έχει πέσει θύμα απαγωγής απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προηγούμενη συνάδελφός μου, η Φερέρο Βάλνερ, είχε δηλώσει επίσημα ήδη από τις 15 Ιουλίου του 2006, δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψή του, ότι πρέπει να απελευθερωθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια της τελευταίας συνάντησης σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου με το Ισραήλ και το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από αυτούς που κρατούν τον κύριο Σαλίτ να τον απελευθερώσουν χωρίς καθυστέρηση. Και συμφωνούμε λοιπόν με την έκκληση και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα. Αυτά τα οποία λέμε συμφωνούν με αυτά τα οποία λένε και οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η σύλληψη και η κράτηση του Σαλίτ είναι αντίθετη με, ε, τα διεθνή, με τους διεθνείς κανόνες. Πρέπει λοιπόν να επιτραπούν και αντιπροσωπείες του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού να τον επισκεφτούν. Γνωρίζω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διαμεσολάβηση για την απελευθέρωση του Γκυλάτ Σαλίτ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς και ελπίζουμε να στεφθούν από επιτυχία. Και εγώ θα ήθελα προσωπικά να πω ότι θα περάσω το μήνυμά σας στην συνάδελφο Κάθη Άστον. Και δεν αγνοώ εδώ επίσης και την οικογένεια του Γκυλάτ Σαλίτ. Ξέρω ότι ο πατέρας του ήταν αυτή την εβδομάδα ανάμεσά της και από ό,τι μαθαίνω αυτή τη στιγμή κάθεται στα έδρανα, στα θεωρία. Θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι οι σκέψεις μας και οι προσπάθειές μας ε, είναι μαζί του. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε αυτόν και όλους όσους υποφέρουν από τις συνέπειες αυτής της απαράδεκτης ε, σύγκρουσης. Ευχαριστώ κύριε Ποτόρσνικ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Επτά, όπως είπα, είναι την προτάση ψηφίσματος για τις οποίες θα κάνουμε ψηφοφορία μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Το επόμενο θέμα είναι η κλιμάκωση τη βίας στο Μεξικό. Και θα ακούσουμε